παράγραφος πρώτη του κανονισμού διαβιβάζεται αυτό το αίτημα στην αρμόδια νομική επιτροπή. Στη συνεδρίαση τη 9 η Σεπτεμβρίου 2013 σα ανακοίνωσα ότι ο κύριο Γκαμπριέλε Αλμπερτίνη, πρώην Ευρωβουλευτή, ε, έκανε αίτημα για την προστασία τη κοινοβουλευτική του ασυλία. Ε, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμό, το αίτημα αυτό διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η εν λόγω Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση τη 14 η Οκτωβρίου 2013, 5 η Νοεμβρίου 2013 και εκ νέου στι 10 Φεβρουαρίου 2014 ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Με επιστολή της 11 Φεβρουαρίου 2014 μου διαβίβασε η Επιτροπή ε, την σύσταση να μην επαναληφθεί η διαδικασία για την προστασία της ασυλίας του κυρίου ε, Αλμπερτίνη, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ε, ελέγξουμε και πάλι την απόφαση του Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2013. Τότε είχε αποφασίσει το Κοινοβούλιο να μην προστατεύσει την ασυλία του κυρίου Αλμπερτίνη. Αν δεν διαφωνείτε, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 9 του κανονισμού θα διαβιβάσω